Καλησπέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Αρχίζουμε και την ε, συνεδρίαση της Επιτροπής μας. Πρώτα απ' όλα να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη παρακαλώ. Εφόσον ε, δεν υπάρχουν αλλαγές, εγκρίνεται. Σημείο 2. Ανακοινώσεις της Πρόεδρου. Στις 16 Οκτωβρίου οι συντονιστές αποφάσισαν να να θέσουν νομοθετική γνωμοδότηση για την οδηγία όσον αφορά την ισορροπία επαγγελματική και προσωπική ζωή στο ΕΛΚ. Να συντάξουν επίση έκθεση στρατηγική σημασία για το πακέτο πάλι ισορροπία επαγγελματική προσωπική ζωή, ώστε ευρωπαϊκά κονδύλια να βοηθήσουν στην ισορροπία αυτή. Ανατέθηκε στο ΕΛΚ να συντάξουν γνωμοδότηση στην έκθεση πρωτοβουλία της Επιτροπής Πολιτισμού για τον εξυγχρονισμό της εκπαίδευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ανατέθηκε στο ΕΛΚ. Επίσης, να αναθέσει δύο γνωμοδότησεις για το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα για την Ισότητα το είναι κάτι που ανέθεσε για τον προϋπολογισμό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επιτροπή μας ΦΑΜ και εμείς το αναθέτουμε στην εισηγήτρια για τον προϋπολογισμό του 2018 της Επιτροπής μας, την κυρία Ματέρα. Επίσης, σύνταξη ε, έκθεση όσον αφορά για το συντονισμό την ε, ετήσια ανάπτυξη 2018 και αποφασίστηκε να ανατεθεί στους σοσιαλιστές. Να συνταχθεί επίσης γνωμοδότηση για ε, έκθεση πρωτοβουλίας της ε, ΛΥΜΠΕ και να ανατεθεί η γνωμοδότηση αυτή στους σοσιαλιστές. Επίσης, να συντάξουμε προφορική ερώτηση με ψήφισμα όσον αφορά τον ακροτηριασμό γενετικών οργάνων εν ώψη της Συνόδου του Φεβρουαρίου, όπου θα έχουμε την Διεθνή ημέρα για μηδενική ανοχή στην κλητοριδεκτομή. Αυτά για το Φεβρουάριο του 2018. Επίσης, όσον αφορά την κατάρτιση του προϋπολογισμού με γνώμονα το φύλλο, επίσης αποφασίσαμε να συντάξουμε γνωμοδότηση και ζητήσαμε επίσης την ε, Επιτροπή Πολιτικής να μας βοηθήσει στην ε, σύνταξη σχετικής έκθεσης. Επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη. Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Δύο Φύλων. Προχωρούμε σημειωτών. Η παρουσίαση θα γίνει από την Βεργίνια Λάγκμπακ, με την οποία θα ανταλλάξουμε απόψεις. Οπότε, παρακαλώ, έχετε το λόγο, κυρία Λάγκμπακ. Σας ευχαριστώ πολύ και είμαι πολύ ευτυχής γιατί τρεις εβδομάδες ε, αφότου ξεκινήσαμε στο Συμβούλιο με το θέμα αυτό έχουμε διαπιστώσει ότι όσοι ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα της ισότητας επικεντρώνονται και πάλι στο θέμα του δίκτυ. Έχουμε λοιπόν μια έκθεση να δώσω στη δείχνω όσοι έχετε χρόνο στην υπηρεσία δημοσιεύσεων υπάρχει μεγαλύτερη έκθεση με πολύ περισσότερα στοιχεία όσον αφορά τον δίκτυ για να ενημερωθείτε. Τώρα με αυτή τη μικρή έκθεση έχετε μια σύντομη ενημέρωση για τον δίκτυ αυτό. Ποια είναι τώρα τα κύρια στοιχεία. Είναι πολύ σημαντικό, ίσως να μην είχατε όλη την ευκαιρία να γνωρίσετε το δίκτυ αυτό, αλλά σας δείχνουμε ποιοι μας στηρίζουν κατά διάρκεια εκπόνησης αυτού του δίκτυ, αλλά και άλλων. Είναι ένα συλλογικό έργο, λοιπόν, όλοι αυτοί οι φορείς μας στηρίζουν το Ίδρυμά μας. Είναι επίσης πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι ο δείκτης ισότητας μεταξύ των δύο φύλων του Ευρωπαϊκού Στιτούτου για την Ισότητα των Δύο Φύλων είναι κάτι για την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο. Οπότε διαπιστώνονται διαφορές μεταξύ των διαφόρων δικτών που κυκλοφορούν στον κόσμο και ο λόγος είναι ακριβώς αυτός, ότι εμείς εξετάζουμε τι ισχύει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τι απορρέει από τις ευρωπαϊκές πολιτικές και εκπονούμε τέτοιους δείκτες για να μπορέσουμε να συγκρίνουμε 28 χώρες μέλη για τα θέματα ε, τα οποία έτσι καλώς μετρούμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι καλό που διαπιστώνουμε ότι τώρα αποτελούμε σημείο αναφοράς όλο και περισσότερο. Είναι ένα δείκτης ο οποίος περνάει τώρα και στο θέμα της ε, πολιτικής που το χρησιμοποιούν οι πολιτικοί. Άλλος λόγος που υπάρχουν διαφορές με τους άλλους δείκτε που κυκλοφορούν είναι ότι εδώ μετρούμε τη διαφορά μεταξύ ανδρών και γυναικών. Δεν μετράμε πόσα σχολεία, για παράδειγμα, έχει για κορίτσια μια χώρα και πόσα για αγόρια. Όχι, εμείς μετρούμε πως οι ίδιες πολιτικές οι οποίες έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε τι διαφορετικό αποτέλεσμα οδηγούν για τους άντρες και τις γυναίκες που ζουν στη μία ή την άλλη χώρα ή στην ίδια χώρα, αν διαπιστώσουμε ότι άλλο είναι το αποτέλεσμα για τα αγόρια και άλλο για τα κορίτσια. Έχουμε από το 0 μέχρι το 100. Θα δείτε κάποιες διαφάνειες όπου θα δείτε ότι οι χώρες που έχουν χαμηλές επιδόσεις σημαίνει ότι έχουν μεγάλες διαφορές ότι είναι μεγάλη η διαφορά μεταξύ αντρών και γυναικών και δεν δείχνουμε αν είναι κάτι αρνητικό για τις γυναίκες ή για τους άντρες. Μόνο όταν αναλύσουμε τα δεδομένα βλέπουμε αν η αρνητική τάση είναι για τους άντρες. Βέβαια, στατιστικά έχουμε διαπιστώσει ότι τις περισσότερες φορές τα αρνητικά δεδομένα είναι για τις γυναίκες. Έπειτα έχουμε και τα επίπεδα επιδόσεων. Αν έχετε πολύ κακή ανάπτυξη στη μία χώρα και είναι εξίσου κακή για τους άντρες και τις γυναίκες, τότε έχουμε και έναν συντελεστή ο οποίος βοηθάει να εκφράσουμε τα τελικά αποτελέσματα. Γιατί δεν μπορούμε να συγκρίνουμε μια χώρα που έχει συνολικά κακά αποτελέσματα με μια χώρα η οποία έχει καλά αποτελέσματα συνολικά χρειάζεται να γίνει μια διόρθωση και χρησιμοποιούμε ένα συντελεστή για αυτήν την διόρθωση ακριβώς. Να λοιπόν τι τομείς εξετάζουμε. 20-21 Νοεμβρίου η πρόεδρος της Επιτροπής σας θα το επιβεβαιώσει θα ξεκινήσουμε μαζί με έναν τομέα του δίκτυα αυτού εδώ στο Κοινοβούλιο θα κάνουμε την παρουσίαση και πρόκειται για την βία σε βάρος των γυναικών. Ε, πρόκειται για ένα δορυφορικό domain και δεν πρόκειται να σας πω τώρα πολλά, γιατί έχουμε ακόμα σχεδόν δύο εβδομάδες μέχρι εκείνη τη στιγμή. Πάντως αυτό το οποίο εμείς βλέπουμε και πώς βλέπουμε εμείς την ανισότητα μεταξύ των δύο φίλων λέμε ότι και η βία σε βάρος των γυναικών απορρέει από την ανισότητα αυτή και ότι η ανισότητα είναι η αιτία της βίας σε βάρος των γυναικών και είναι κάτι που συζητούμε με διάφορους εμπειρογνώμονες. Εμείς δεν έχουμε βάλει την βία σε βάρος των γυναικών σαν ένα κεντρικό στοιχείο του δίκτυ, αλλά πρέπει με κάποιο τρόπο να εξετάσουμε και το θέμα της βίας σε βάρος των γυναικών. Το κομμάτι που είναι έτσι πορτοκαλό καφέ είναι ένα καινούριο, το οποίο εκτίμησαν πάρα πολύ. Ότι δηλαδή εξετάζουμε και την διασύνδεση μεταξύ των ε, διαφόρων ε, ανισοτήτων. Είναι αυτό που το λέμε intersecting inequalities, ο κύκλος γύρω-γύρω από όλα τα μικρά κυκλάκια γιατί δεν φτάνει να δούμε το δίκτυο όσον αφορά τη γνώση, το χρόνο, την υγεία κτλ. Οι άντρε μεταξύ του διαφορετικοί, οι γυναίκε είναι διαφορετικέ, οπότε προσπαθήσαμε να πάρουμε πολλά στοιχεία μαζί. Την ηλικία, την αναπηρία, την εκπαίδευση, το τύπο οικογένειας. Και όσο είχαμε στοιχεία στην, περισσότερα στη διάθεσή μας, φαίνεται και στην έκθεσή μας αυτή εδώ, ε, διαπιστώνουμε πόσο μεγάλες μπορεί να είναι οι διαφορές για άντρες και γυναίκες ε, που είναι ανάπηροι ή μεταξύ αντρών και γυναικών που έχουν τα ίδια επίπεδα γνώσης. Είναι πολύ σημαντικό να διαπιστώσουμε και να μελετήσουμε ποιες είναι οι διαφορές μέσα στην κάθε ομάδα που εξετάζουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, εξετάζουμε το τομέα της εξουσίας, της ισχύω. Εδώ έχουμε μεγάλη βελτίωση σε κάποιες χώρες. Πρώτη, πρώτο έπαθλο, η Ιταλία, σε σχέση με πριν από 10 χρόνια. Είχε την μεγαλύτερη βελτίωση και γενικά στον δίχτυ, όχι μόνο στον τομέα της εξουσίας. Ιταλία, μετά έρχεται η Γαλλία και μετά η Σλοβενία. Έχουν βελτιώσει δηλαδή πολύ μέχρι το 2012 την κατάσταση. Και εδώ βλέπουμε και ποιε είναι αυτές οι χώρες οι οποίες αντί να πάνε μπροστά πήγαν πίσω. Η Φιλανδία, η Σλοβακία και η Τσεχία. Η Φιλανδία και η Τσεχία οπισθοχώρησαν και από το 2012 και μετά. Και βέβαια οι χώρες πρέπει να δούνε γιατί. Και εδώ δεν πρόκειται μόνο για την πολιτική εξουσία, έτσι. Τώρα εισάγουμε και άλλους δείκτες για να εξετάσουμε τα ποσοστά γυναικών και ανδρών σε διάφορες ερευνητικές οργανώσεις, στον αθλητισμό, έρευνα, αθλητισμό και ξέχασα τα υπόλοιπα το τρίτο. Οπότε έχουμε και νέους δείκτες για να δούμε τι γίνεται και με την κοινωνική εξουσία. Ποιες είναι οι κυριότερες διαφορές στις διάφορες χώρες μεταξύ αντρών και γυναικών. Ο ιδιωτικός τομέας βέβαια προχωράει ε, ολοταχώς όσον αφορά το θέμα της εξουσίας. Εδώ βλέπετε τις χώρες, τις διάφορες χώρες η Σουηδία, η Γαλλία και η Φιλανδία βρίσκονται πάνω-πάνω με τα καλύτερα αποτελέσματα. Η Ουγγαρία, η Ελλάδα και η Τσεχία πρέπει να βελτιώσουν κατά πολύ την κατάσταση. Βλέπετε λοιπόν ότι ναι μεν έχουν μειωθεί τα χάσματα όσον αφορά την εξουσία, παρόλα αυτά ο δείχτης είναι πολύ χαμηλός πράγμα το οποίο δείχνει ότι στο θέμα της εξουσίας οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών παραμένουν πολύ μεγάλες. Και αν δούμε και τις αποφάσεις τις οικονομικές που λαμβάνονται, διαπιστώνουμε πόσες γυναίκες είναι επικεφαλής κεντρικών τραπεζών. Μόνο 3% υπήρχε βελτίωση τα τελευταία 10 χρόνια. Ε, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής ε, Κεντρικής Τράπεζας ποτέ δεν ήταν οι γυναίκες πάνω από το 10% εκεί. Ή το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Ε, διαπιστώνουμε επίσης ότι στις διάφορες χώρες μέλη οι διοικητές των τραπεζών είναι άντρες, δεν είναι γυναίκες. Η κατανομή λοιπόν εξακολουθεί να επιδέχεται πολλές βελτιώσεις. Η έκθεση τα δείχνει αυτά. Θα βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες εκεί. Έρχομαι τώρα στο θέμα της γνώσης. Εδώ είχαμε μια μικρή βελτίωση κυρίως εξαιτία της ε, εκπαίδευσης, της μόρφωσης. Οι χώρες που βελτιώθηκαν ε, περισσότερο είναι η Λετωνία, η Τσεχή, η Ισπανία, ενώ χειρότερες η Βουλγαρία, η Σλοβακία και το Βέλιο. Λέει η ομιλήτρια, αλλά δεν αναφέρει τα ποσοστά της ε, γνώσης. Εδώ βλέπουμε ότι η μεγαλύτερη πρόκληση σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της γνώσης είναι ότι υπάρχει διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών στην εκπαίδευση. Και αν δείτε τι γίνεται στο τομέα της ευημερίας, διαπιστώνετε ότι αν δεν πληρωνόσαστε αρκετά. Τα τρία τέταρτα είναι γυναίκες. Ενώ αν πάμε στη τεχνολογία, τα μαθηματικά, ε, μηχανική που είναι τα επαγγέλματα του μέλλοντος και πληρώνονται πιο πολύ, εκεί θα διαπιστώσετε ότι κυριαρχούν οι άντρες. Κοιτάξαμε επίσης τι γίνεται και με τη διαβίου ε, μόρφωση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για άτομα χαμηλότερης μόρφωσης. Οι μετανάστες που δεν έχουν ευκαιρίες και αν δεν έχει κανείς περάσει από την επίσημη εκπαίδευση, προφανώς έχει λιγότερες επιλογές στη διάθεσή του. Εδώ λοιπόν βλέπετε τις επιδόσεις των διαφόρων χωρών και οι τρεις καλύτερες είναι οι συνηθισμένες χώρες. Αν δούμε τώρα τον τομέα του χρόνου, τι γίνεται με το χρόνο. Ο χρόνος είναι ο μόνος τομέας στον οποίο δεν βλέπουμε βελτίωση, αλλά επιδείνωση. Αν οι γυναίκες και οι άντρες δουλεύανε μία ώρα παραπάνω για να βοηθούν στο σπίτι, να φροντίζουν τους ηλικιωμένους, τα παιδιά. Τώρα φαίνεται ότι οι άντρες προσφέρουν λιγότερο χρόνο σε αυτά από ό,τι πριν από 10 χρόνια. Αν κοιτάξουμε πού υπάρχει βελτίωση για αυτήν την ε, μη πληρωμένη εργασία, είναι η Λετωνία, η Τσεχία και η Ισπανία. Αλλά αυτοί που βελτιώθηκαν λιγότερο είναι η Βουλγαρία, η Σλοβακία και το Βέλγιο. Σε 12 χώρες μέλη, σε αυτό το τομέα που είναι τόσο σημαντικό για τη ζωή, την καθημερινή, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει επιδείνωση. Εδώ βλέπετε ποια είναι η κατάσταση των διαφόρων χωρών. Η Σουηδία, οι κάτω χώρε και η Δανία βρίσκονται στην καλύτερη κατάσταση. Και εκεί που δεν κατανέμεται καθόλου ισότιμο χρόνο είναι στη Βουλγαρία, την Ελλάδα και τη Σλοβακία. Και εκεί βλέπουμε ότι μόνο το 1 τρίτο των ανδρών καθημερινά ασχολούνται με τα παιδιά, με το νοικοκυριό, με το μαγείρεμα. Τα δύο τρίτα των ανδρών δεν ασχολούνται με αυτό καθόλου. Κάτι το οποίο επίση σημαίνει ότι το βάρος πέφτει στις γυναίκες. Και το αποτέλεσμα είναι ότι οι άντρες... Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουν και ελεύθερο χρόνο. Και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Ο ελεύθερος χρόνος για να ασχοληθούν ίσως με μια κατάρτιση ή με κάτι άλλο που θα θέλανε. Εδώ τώρα ερχόμαστε σε κάποια άλλη ανισότητα όπου συμπεριλαμβάνουμε περισσότερους από αναπαράγοντες. Έχει να κάνει με την καθημερινή φροντίδα. Όταν ζουν μόνοι τους άντρες και γυναίκες, η διαφορά μεταξύ τους δεν είναι τόσο μεγάλη. Στα ζευγάρια που δεν έχουν παιδιά, ούτε και εκεί είναι πολύ μεγάλη διαφορά. Αλλά στην περίπτωση των ζευγαριών με παιδιά, η διαφορά είναι πολύ μεγάλη ή σε μονογονικές οικογένειες. Είναι πολύ ευάλωτες ε, οι γυναίκες αυτές τις περιπτώσεις. Αν λοιπόν είσαστε μητέρα, έχετε τρία παιδιά, για παράδειγμα, τότε είναι πολύ μεγάλη διαφορά σε βάρος της γυναίκας και στην περίπτωση μονογονικών οικογενειών ε, και εκεί υποφέρουν περισσότερο οι γυναίκες. Τώρα να περάσουμε στο θέμα της εργασίας, που κατά κάποιο τρόπο είναι μια από τις βασικές προϋποθέσεις για την ε, οικονομική ανεξαρτησία προκειμένου να μπορεί να κατοχυρώσει συνταξιδοτικά δικαιώματα κάποιος. Αν δούμε εδώ ποιες είναι οι χώρες οι οποίες βελτίωσαν περισσότερο την κατάστασή τους και ποιες την ε, βελτίωσαν λιγότερο. Στην καλύτερη περίπτωση έχουμε τη Μάλτα, το Λουξεμβούργο και την Κύπρο που είχαν περισσότερες βελτιώσεις και λιγότερες βελτιώσεις διαπιστώνουμε στην περίπτωση της Δανίας, της Σλοβακίας και της Ρουμανίας. Από το 2005 όταν κάναμε την ανάλυση η βελτίωση είναι 1,5% συνολικά. Γι' αυτό μιλάμε για αριθμό σημειωτών, ότι πηγαίνουμε πάρα πολύ αργά. Αν συμβαίνουν τόσα πολλά πράγματα και σε 10 χρόνια η βελτίωση είναι μόνο της τάξης του 1,5% καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ μικρή. Εμείς μετράμε βέβαια την πλήρη απασχόληση εδώ στον δίκτυ μας, έτσι, γιατί αλλιώς αν μιλάμε για την μερική απασχόληση τα πράγματα διαφέρουν. Τι σημαίνει Άλλο θα δουλεύει 12 ώρε, άλλο θα δουλεύει 30 ώρε δεν το έχουμε λάβει αυτό υπόψη μα. Μιλάμε για πλήρη απασχόληση. Και τα καλύτερα αποτελέσματα έχουν η Σουηδία, η Δανία και οι κάτω χώρες. Και οι χώρες οι οποίες χρειάζονται βελτίωση είναι η Ιταλία, η Ελλάδα και η Σλοβακία. Και σε πέντε χώρες μέλη διαπιστώσαμε ότι στα δέκα χρόνια δεν υπήρξε καμία αλλαγή. Η ίδια κατάσταση. Η διαφορά λοιπόν στην πλήρη απασχόληση για τις γυναίκες είναι 40 40% των γυναικών έχουν πλήρη απασχόληση, ενώ το 66% των ανδρών. Και αν δούμε και τις γυναίκες με αναπηρίες, τότε και εκεί υπάρχουν πολύ μεγάλες διαφορές. Οι γυναίκες με αναπηρία, μόνο το 19% αυτών δουλεύουν με πλήρη απασχόληση ενώ 28% των ανδρών με αναπηρίες έχουν πλήρη απασχόληση. Αν δούμε τις γυναίκες με χαμηλή μόρφωση, με χαμηλά προσόντα, 17% έχουν πλήρη απασχόληση από αυτές, ενώ πάνω από 30% οι αντίστοιχοι άντρες. Και οι γυναίκες πριν τη συνταξιοδότηση, ηλικία 50 με 60, όσο είμαι και εγώ, μόνο τα 4% των γυναικών αυτών έχουν πλήρη απασχόληση. Διαφορά είναι 19% με τους άντρες. Όταν μιλάμε λοιπόν τώρα για την ασφάλεια, για τα κοινωνικά δικαιώματα, για την προστασία και όλα αυτά τα μέτρα τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τον άνθρωπο να ανταποκριθεί στις αλλαγές. Η ο δείχτης αυτός είναι πολύ σημαντικός για να δούμε τι είναι τελικά αυτό το οποίο λείπει. Στην απασχόληση κάτι άλλο είναι οι διακρίσεις μεταξύ των δύο φύλων. Όπως συμβαίνει και στην εκπαίδευση. Οι περισσότερες γυναίκες στην εκπαίδευση, υγεία από τη μία και από την άλλη μεριά έχουμε τις τεχνολογίες που έχουμε περισσότερους άντρες. Στην εκπαίδευση έχουμε περισσότερες γυναίκες. Δεν αλλάζει αυτό. Υπάρχει λοιπόν διάκριση στην απασχόληση και αυτή η διάκριση αντιστέκεται. Οχτώ στους δέκα είναι άντρες στη τεχνολογία ενώ το αντίστοιχο ποσοστά για τις γυναίκες είναι στον τομέα της φροντίδας και της εκπαίδευσης. Εδώ βλέπουμε ποιες ομάδες είναι περισσότερο εκτεθειμένες στη διάκριση αυτή. Και πάλι είναι οι μονογονικές οικογένειες και τα ζευγάρια με παιδιά. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να δουλέψει κανείς με πλήρη απασχόληση σε αυτές τις περιπτώσεις. οι διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι 28% στα ζευγάρια με παιδιά, που είναι πολύ μεγάλη για να την αγνοήσουμε. Γιατί μας δείχνει πού πρέπει να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας. Έρχομαι τώρα στο χρήμα. Εδώ έχουμε τις χώρες που βελτίωσαν την κατάσταση και αυτές που δεν την βελτίωσαν τόσο. Βλέπετε εδώ ποιες είναι αυτές. Τα χρήματα μας ε, εξασφαλίζουν και τη ζωή και την αξιοπρέπεια που θέλουμε. Είδαμε ότι οι γυναίκες μορφώνονται λιγότερο Αν έχεις χρήματα, μπορείς να κάνεις και κάποια αποταμίευση και να μπορέσεις έτσι να καλύψεις κάποιες από τις διαφορές με το άλλο φύλλο. Στα κέρδη η διαφορά είναι δύο φορές μεγαλύτερη στα ζευγάρια με παιδιά. Στην περίπτωση δηλαδή που έχουμε ε, ζευγάρια με παιδιά ή μονογονικές οικογένειες, τα μισά τελικά βγάζει η γυναίκα από τον άντρα. Και το 75% κινδυνεύουν από φτώχεια. Και η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη, δύο φορές χειρότερη, αν δεν έχουν γεννηθεί μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι Πολύ σημαντικό λοιπόν να μην ξεχνάμε αυτόν τον παράγοντα. Και τώρα έρχομαι στο συνολικό δίκτυ και τα αποτελέσματα. Τι βλέπουμε λοιπόν εδώ. Βλέπουμε ότι οι καλύτερες επιδόσεις είναι της Ιταλίας 12,9% βελτιώθηκε Έκανε πολλά και μπορεί να είναι περήφανη η Ιταλία για τα αποτελέσματα. Και η δεύτερη καλύτερη χώρα είναι η Κύπρος και μετά είναι η Σλοβενία και η Ιρλανδία. Τώρα αυτές που βελτιώθηκαν λιγότερο σε, όλα, σε όλους αυτούς τους τομείς έτσι, είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Τσεχία και η Σλοβακία που δεν είχαμε σχεδόν καμία διαφορά. Πολλές ε, χώρες βελτιώθηκαν σε πολλούς τομείς, αυτά μπορείτε να τα διαβάσετε στην ε, έκθεση. Και αν δούμε συνολικά το σκορ για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ έχετε ενταξινόμηση των χωρών. Σε 10 χρόνια, λοιπόν, τέσσερις βελτίωσαν την κατάστασή τους. Γι' αυτό και μιλάμε για πολύ αργό ρυθμό φιδιού. Τέσσερις μονάδες σε 10 χρόνια, αν λάβουμε υπόψη μας όλα έχουμε κάνει και όσες προσπάθειες έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση που θέλει να είναι παράδειγμα στον κόσμο. Ε, λοιπόν και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολλά μένει να γίνουν. Η Σουηδία, η Δανία είναι οι δύο καλύτερες, η Φιλανδία 100 χώρες ακολουθούν. Ήταν πάντα έτσι κι αλλιώς όλους τους δείχτες λίγο πολύ καλύτερες. Και από την άλλη μεριά η Ελλάδα είναι στη χειρότερη θέση. Η Ουγγαρία μετά, η Σλοβακία ακολουθούν και μιλάμε για πρόοδο. Πρέπει συστηματικά να προσπαθήσουμε να πάρουμε τα μέτρα που χρειάζεται και να τα εφαρμόσουμε. Η εξουσία, η γνώση και ο χρόνος είναι αυτά που κυριαρχούν. Και όταν μιλάμε για εξουσία, Ας δούμε τι γίνεται στη Γερμανία, για παράδειγμα, μέσω της νομοθεσίας, συζητήσεων. Είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για να αλλάξει η κατάσταση. Για να καλυφθεί αυτό το μεγάλο χάσμα που έχουμε στην ε, εξέλιξη της εξουσίας στα χέρια των ανδρών και των γυναικών. Επίσης, οι διακρίσεις μεταξύ των δύο φύλων που οδηγεί στις διαφορές των συντάξεων, το τι υποβαθμίζεται η απασχόληση των γυναικών, όλα αυτά είναι προκλήσεις που πρέπει να συζητηθούν. Όπως επίσης τα στερεότυπα, η εκπαίδευση, η κατάρτιση. Πρέπει να αλλάξει αυτή η διάκριση μεταξύ ανδρών και γυναικών στην απασχόληση. Και φυσικά το θέμα του καταμερισμού του χρόνου δεν είναι κάτι που πρέπει να καθόμαστε και να κοιτάμε, κάτι πρέπει να κάνουμε, γιατί είναι πολύ άνηση η κατάσταση. Πρέπει να βοηθήσουμε τις γυναίκες λοιπόν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο γενικά, αλλά και πολύ συγκεκριμένα. Ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε, κυρία Λάμπεκ, ε, για την παρουσίαση της ε, κατάστασης στα διάφορα κράτη-μέλη. Ο δείκτης ισότητας των φύλων ε, μας βοηθάει πολύ να καταλάβουμε καλύτερα την κατάσταση, ποιες αλλαγές έχουν γίνει, ποιες δεν έχουν γίνει. Τώρα θα δώσω <clears throat> το λόγο στα μέλη, Κυρία κυρία είναι, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω το ΕΙΓΕ για την παρουσίαση του δίκτυα αυτού. Γιατί πολύ συχνά αυτό που δεν μπορούμε να δούμε δεν μπορούμε και να το διορθώσουμε, γιατί θεωρούμε ότι δεν υφίσταται. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να είμαστε πολύ υποστηρικτικοί και υπό την έννοια των πόρων προς το έγκαιο για να συνεχίσει με τη δουλειά αυτή. Αφενός αυτό. Αφετέρου, αναρωτιέμαι αν θέλαμε να έχουμε αυτές τις ε, παρουσιάσεις ε, τις κυλιόμενες πλησιάζοντας τι εκλογές σε διάφορα κάτι μέλη ώστε το έγκυ να παρουσιάσει τα αποτελέσματα αυτά και να μπορέσουμε να συναντήσουμε τα τοπικά μέλη των ε, κοινοβουλίων και άλλους φορείς για να συζητήσουμε ποια, πώς έχει η κατάσταση εκεί. Και κάτι που βέβαια δεν είναι νέα, αλλά είναι ανησυχητικό, είναι αυτή, αυτός ο ρυθμός χελώνας. Δηλαδή ότι η όποια βελτίωση, η όποια αλλαγή δεν έρχεται ταχαίως. Και έχουμε και οικονομικές διαφορές έχουμε και διαφορές ρυ, ρυθμιστικές και είναι σημαντικό να αναλάβουμε τις δράσεις που πρέπει να αναλάβουμε. Γιατί συζητούμε για κάποιες ρυθμιστικές πράξεις ή ποσοστώσεις και λέμε πάντοτε θα προσπαθήσουμε πρώτα τις, τα εθελοντικά μέτρα. Και απλώς με την ενημέρωση, με την ευαισθητοποίηση ελπίζουμε ότι τα προβλήματα θα επιληθούν. Το δύσκολο λοιπόν μάθημα προκύπτει από την ιστορία ότι, ότι δεν συμβαίνει αυτό. Χρειάζονται δεκάδες και εκατοντάδες τελικά χρόνια για να βελτιωθούν τα πράγματα αυτά έτσι από μόνα τους. θα ήθελα αυτό να το συνδέσω μάλιστα με κάτι άλλο που θα συζητήσουμε εδώ. Το σχέδιο δράσεως για την ισότητα των φύλων. Τι προτείνουμε στα πλαίσια του σχεδίου αυτού. Νομίζω ότι στο μέλλον αυτό που θα χρειαστούμε για αυτό το σχέδιο δράσεως είναι μία ποσοτική καταμέτρηση, συγκριτική αξιολόγηση του τι μπορούμε να κάνουμε και χρειαζόμαστε επίσης και ανάληψη διορθωτικής δράσης. Γιατί θα πρέπει να είναι υπεύθυνα τα κράτη-μέλη και οι υπόλοιποι φορείς για τις επιδόσεις τους. Αν δεν βλέπουμε αποτελέσματα από τα διάφορα σχέδια δράσης σε επίπεδο κάτους μέλους, για την ισορροπία της οικογενειακής ε, και επαγγελματικής ζωής και τα λοιπά, Τότε τι πρέπει να γίνει με τα συγκεκριμένα αυτά ζητήματα που εκκρεμούν. Και ίσως θα μπορούσαμε να αναλάβουμε πιο ισχυρή δράση. Δηλαδή κατόπιν μιας τέτοιας μελέτης θα μπορούσαμε να κάνουμε μια συγκριτική αξιολόγηση των δικτών αυτών που έχουμε αναχώρα με τους στόχους σχεδίου δράσεως ώστε να μπορέσουμε να αναλάβουμε διορθωτικές δράσεις και αν δεν υπάρξει βελτίωση θα πρέπει να βγει το συμπέρασμα ότι αυτές οι διορθωτικές δράσεις δεν είναι επαρκείς. Και νομίζω ότι θα άξιζε τον κόπο αυτές οι κυλιόμενες συζητήσεις και επαφές με τα τοπικά μέλη των κοινοβουλίων να συνεχίζονται για 5-10 χρόνια. Να έχουμε ένα βάθος δηλαδή. Και μέσω αυτής της κριτικής αξιολόγησης να προσπαθούμε να διευρύνουμε δίκτυα και συμμαχίες με τα τοπικά μέλη των κοινοβουλίων για να αυτά τα ζητήματα. Βεβαίως έχουμε και νέα θέματα που σχετίζονται με την ψηφιοποίηση, με τις πολλαπλές διακρίσεις, με ανθρώπους που εργάζονται στο εξωτερικό, με τα συνταξιοδοτικά. Τώρα εντάξει, δεν θα τα καταλογοποιήσω γιατί χρειαζόμαστε και πόρους για να δούμε όλες αυτές τις υπόλοιπες περιοχές, αλλά σε ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ. Η κυρία Ward έχει το λόγο, λέει πρόεδρος. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Εμείς ε, εκτιμούμε τις ενδείξεις αυτές, τα στοιχεία αυτά που συλλέγεται όταν μπορούμε μάλιστα να τα χρησιμοποιήσουμε και στη δουλειά μας, στις δικές μας μελέτες. Ήθελα δύο στοιχεία να αναφέρω. Καταρχάς, φαίνεται ότι τα τελευταία δέκα χρόνια δεν έχει σημειωθεί ουσιαστικά πρόοδος. Ε, χρόνια στα οποία είχαμε την κρίση και είχαμε και πολλά λιτότητα λιτότητας από πάρα πολλά κράτη-μέλη. Εγώ είμαι βέβαιη ότι οι γυναίκες είναι αυτές που σήκωσαν το βάρος της λιτότητας στην πραγματικότητα. Και το βλέπουμε αυτό χαρακτηριστικά στην κατανομή του χρόνου. Δεν έχουν πλέον χρόνο οι γυναίκες. Και όταν μιλάω με ομάδες, με ενώσεις γυναικών, ακούω ότι πάρα πολλές από αυτές πρέπει να έχουν πολλές δουλειές για να μπορούν απλώς να πληρώνουν το λογαριασμό. Ήμουν σκιώδης και στην έκθεση για τους στόχους κατά της στόχιας και το αυξανόμενο κόστος των οικοκυριών και είχαμε υπογραμμίσει ότι προκειμένου τα νοικοκυριά να μπορούν να πληρώνουν το κόστος, το λογαριασμό της θέρμανσης του ηλεκτρικού κτλ. Πρέπει οι γυναίκες να δουλεύουν όλο και περισσότερο απλώς και μόνο, όχι για να έχουν περισσότερα χρήματα για διακοπές και λούσα, αλλά για να μπορούν να πληρώνουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Επομένως, στην κατανομή του χρόνου φαίνεται ξεκάθαρα ότι δεν έχει σημειωθεί πρόοδος την ίδια στιγμή που τα μέτρα λιτότητας επιβλήθηκαν. Την ίδια περίοδο δηλαδή. Η επίσκεψή σας εδώ μας βρίσκει σε μια στιγμή όπου είναι στο προσκήνιο η βία που ασκείται στις γυναίκες, η παρενόχληση, η εκμετάλλευση, όλα αυτά γνωρίζουμε ότι συμβαίνουν πάρα πολύ καιρό, πάρα πολλά χρόνια. Τα σκάνδαλα της στιγμής θα συνεχιστούν βεβαίως, γιατί τώρα έχει ανοίξει το θέμα, όχι μόνο στις τέχνες και στα θεάματα, αλλά και στο πολιτικό πεδίο και από διάφορες ε, ε, επαγγελματικές ε, θα τίθεται το θέμα άλλο και περισσότερο. Αναρωτιέμαι λοιπόν στη συλλογή των δεδομένων σας με τα συμπεράσματα που εσείς βγάζετε πώς θα μπορούσαμε καλύτερα να καταδείξουμε το πρόβλημα που έχουμε. Γιατί για μένα είναι σαφές. Όταν οι γυναίκε δεν είναι εμφανεί ω μέλη της κοινωνίας τότε είναι πιο εύκολο να αντισκεφτεί ως αντικείμενα να τις εκμεταλλευτεί κανείς πιο εύκολα δηλαδή. Και είναι πιο εύκολο να υπάρχουν αυτά τα ανοίγματα, αυτή η παρενόχληση σεξουαλική και άλλη προς τις γυναίκες. Πώς μπορούμε λοιπόν να καταδείξουμε, να δείξουμε την ανάγκη της αλλαγής ισορροπίας στην εξουσία γιατί αν δεν έχουμε περισσότερες επιφανείς και εμφανείς γυναίκες θα συνεχιστούν όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γκέρεκε, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ για την έκθεση αυτή, για την παρουσίαση. Ήταν πολύ ωραίο να λάβουμε μια τόσο πλήρη επισκόπηση. και αναρωτιέμαι σχετικά με τη διάκριση ανάμεσα στις γυναίκες και στις μητέρες, στον ιδιαίτερο ρόλο που έχουν ε, να συνοδεύουν την οικογένειά τους. Και όσον αφορά την αξιολόγηση των διαφόρων ε, χωρών, ε, υπάρχουν και διάφορες υποκατηγορίες. Για παράδειγμα, όσον αφορά την φροντίδα των μελών της οικογένειας. Δεν καταλαβαίνετε τι λέω? Ε, νομίζω ότι είναι σημαντικό να καταλαβαίνετε τι λέω. Όταν μιλάμε για την φροντίδα άλλων ανθρώπων, ε, έχει διαφορά εάν ε, επιτρέπεται η ευθανασία ή η το να συνοδεύσει κανείς σε την ε, διαδικασία προς το θάνατο. Αυτό έχει νομικά διαφορά και επίσης ε, όσον αφορά το εισόδημα, μιλάμε για τα χρήματα, αλλά με ή χωρίς παιδιά, διότι πρέπει να εξετάσουμε και το φορολογικό βάρος. διότι η φορολογία εισοδήματος συνήθως είναι ψηλότερη για όσους δεν έχουν παιδιά. Και δεν ξέρω εάν έχει ληφθεί υπόψη στην ε, έκθεσή σας ε, η περίπτωση όπου αυξάνεται η φορολογία για τους γονείς. Θα πρέπει δηλαδή να δούμε και τις σχέσεις ανάμεσα στα στοιχεία. Γιατί, για παράδειγμα, ένα κράτος βρίσκεται πολύ ψηλά όσον αφορά την φροντίδα των μελών της οικογένειας και το θέμα ε, της φροντίδας ε, όσων πεθαίνουν ή ε, της ευθανασίας και αυτό είναι πολύ σημαντικό. νομίζω ότι μπορείτε να πλουτίσετε έτσι την έκθεση σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ε, η κυρία Σόντροβα, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την μελέτη αυτή και την πολύ σαφή μεθοδολογία που χρησιμοποιεί το Ινστιτούτο σας. Εγώ προσωπικά περιμένω παρακολούθηση όλων των δικτών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ακριβώς κάνετε εσείς και θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει και ανταλλαγή ε, βέλτιστων πρακτικών. Συμφωνώ με τη συνάδελφη Επιτικάινεν ότι είναι απαραίτητο να ε, διαδίδουμε, να δημοσιεύουμε τα αποτελέσματα στα κράτη-μέλη. Πιστεύω ότι πρέπει να δοθεί περισσότερη προσοχή στα αποτελέσματά σας. Αναρωτιέμαι λοιπόν αν το Ινστιτούτο σας οργανώνει διασκέψεις ε, Προσφέρετε να παρουσιάσει τα δεδομένα αυτά στα κράτη-μέλη, διότι είναι πολύ χρήσιμα αυτά που κάνετε. Η συστηματική συνέχιση της ε, διαξαγωγής των ερευνών σας ε, θα ε, βελτιώσει τα διαθέσιμα στοιχεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι έρευνες αυτές μας δείχνουν ότι η κατάσταση γενικά βελτιώνεται. Αυτή είναι η εντύπωσή μου και συμφωνώ ότι δεν θα πρέπει να εφησυχάσουμε όσον αφορά τον ρυθμό. Από την άλλη, ας είμαστε δίκαιοι να εκτιμήσουμε τις προσπάθειες και των ε, κρατών μελών και των μη κυβερνητικών οργανώσεων ε, σε πολλές περιοχές ε, η κατάσταση για τις γυναίκες είναι πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν. Μπορεί όλα αυτά να μην γίνονται με την ταχύτητα που θα θέλαμε, βλέπουμε όμως να σημειώνεται πρόοδος. Για παράδειγμα, όσον αφορά ε, τον τομέα της ε, ισχύω των εξουσιών αναφερθήκατε στις πολύ σημαντικές διαφορές που υπάρχουν και νομίζω ότι στον τομέα αυτών οι πολίτες ε, καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι ναι, μας λείπουν οι γυναίκες ε, στην πολιτική. Ε, συμφωνώ ότι δεν θα προχωρήσουν τα πράγματα από μόνα τους, αλλά και οι ψηφοφόροι μας θέλουν να δουν περισσότερες γυναίκες στις τοπικές αρχές, στο κοινοβούλιο, στα δημοτικά συμβούλια. Γι' αυτό είμαι υπέρ της προώθησης των βέλτιστων πρακτικών ε, και των ε, καλών παραδειγμάτων. Νομίζω ότι πολλοί κόσμος ενδιαφέρεται πολύ για το θέμα αυτό. Και μία ερώτηση. Θα ήθελα πολύ να ακούσω περισσότερα στοιχεία όσον αφορά την οικονομία. Ε, αναφέρατε ότι στην Τσεχία, στη χώρα μου, τα αποτελέσματα είναι μηδενικά. Από την άλλη, είδα και το διάγραμμα όπου νομίζω ότι υπάρχει μια αύξηση της τάξης του 5% από ό,τι μπορούσα να καταλάβω. Κάνω λάθος. Ε, υπήρχε λοιπόν πραγματική πρόοδος, έστω και ελάχιστη. Και όταν αναφέρεστε στις αιτίε που αυξάνεται το χάσμα. Να σας πω τη δική μου άποψη. Νομίζω ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα σε αυτά που ανέφερε η συνάδελφος Έρικα, ο αριθμός των γυναικών που αναλαμβάνουν τη φροντίδα των παιδιών τους ε, αυξάνεται και αυτό έχει αρνητικές συνέπειες στην οικονομία τους. Υπάρχει λοιπόν ε, σχέση ε, ανάμεσα στον αριθμό των γυναικών που παίζουν πιο σημαντικό ε, ρόλο ως μητέρες και στην πιο πολύπλοκη πορεία της σταδιοδρομίας τους. Αλλά δεν θα πρέπει να θεωρήσουμε πάντα ότι αυτό είναι αρνητικό φαινόμενο. Εγώ λοιπόν θα ήθελα να δω αυτό ακριβώς τη σχέση ανάμεσα στις γυναίκες που έχουν γονική άδεια ή και διότι αυτό αυτά τα χρονικά διαστήματα δεν θα πρέπει να θεωρηθούν αρνητικά. Σας ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Λάμπακ. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο στη διάθεσή μας, γιατί στις 4 θα ξεκινήσουμε, την κοινή, θα ξεκινήσουμε λέει, η Πρόεδρος την κοινή συνεδρίαση. Αν μου επιτρέπετε, θα ξεκινήσω από το τελευταίο νομίζω ότι είπα σχεδόν καμία αλλαγή. Το γράφημα σωστό είναι και σωστό είναι και αυτό που είπατε κι εσείς. Τώρα για το συσχετισμό, αυτό που είπατε. Και αυτό ίσως συνδέεται και με το ερώτημα για κάποιες ε, θεσμικές, ίσως ε, επίσημες, εν πάση περιπτώσει, υπηρεσίες για του ανθρώπου που αντιμετωπίζουν κάποια νόσο ή αναπηρία κτλ. Εκεί είναι που χρειάζεται ισχυρό δείκτη. Πρέπει να είναι συγκρίσιμα τα στοιχεία, πρέπει να είναι τακτικά διαθέσιμα, ώστε να μπορούμε να τα εξετάσουμε και να τα συγκρίνουμε. Οι συσχετισμοί που κάνουμε είναι επιπλέον δεν τοποθετούμε όλα αυτά τα στοιχεία στη βαθμολόγηση, γιατί η βαθμολόγηση πρέπει να ακολουθεί την αυστηρή μεθοδολογία, αλλά προσπαθούμε να δώσουμε το πλαίσιο. Όλα αυτά που αναφέρατε είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα και πολύτιμα. Και κάθε φορά που σχεδιάζουμε τη δομή του δίκτυ, τα στοιχεία από τα οποία αντλεί, το επόμενο σχέδιο θα είναι το 19 για την ισορροπία επαγγελματική και προσωπική ζωή. Λαμβάνουμε υπόψη διάφορα στοιχεία λοιπόν και θα μπορούσαμε να λάβουμε και αυτά. Για παράδειγμα, τα θέματα νομοθεσίας δεν ασχολούμαστε με αυτά. Γιατί θεωρούμε πόσο ο κάθε άνθρωπος θεωρεί ο, ο ίδιος ότι ασχολείται, ότι αναλαμβάνει ένα καθήκον χωρίς μισθό, ας πούμε, μη πληρωμένο. Τώρα, για τις κυλιόμενες παρουσιάσεις που παρουσιάσατε, τα road show, έχουμε προετοιμάσει τέτοιες παρουσιάσεις πριν από τα μέσα του επόμενου έτους θα έχουμε δελτία επεξηγηματικά φυλάδια σε όλες τις γλώσσες των κρατών μελών για τις πιο σημαντικές προκλήσεις επισκεπτόμαστε την κρατημέλη και θα μπορούσαμε και με τη δική σας συμμετοχή να έχουμε περισσότερες επισκέψεις και προς τα κοινοβούλια και προς το κοινοβούλιο επίσης το ευρωπαϊκό. Τώρα για το συσχετισμό με την ε, λιτότητα. Νομίζω ότι στον επόμενο σχεδιασμό του δίκτυ θα μπορούσαμε πράγματι να αναπτύξουμε και την πρωτοβουλία για την ε, εξισορρόπηση προσωπικής και επαγγελματικής ζωής και πώς θα μπορούσαν να συνδεθούν οι δείκτες αυτοί και για τα θέματα της, ε, για τα κρούσματα βίας κατά των γυναικών ίσως είναι ενδιαφέρον να ακούσετε ότι πριν από ένα χρόνο περίπου είχαμε αναπτύξει και το δοκιμάζουμε τώρα μια αξιολόγηση για ένα online μέσο που θα κατέγραφε την, το στοιχείο της ισότητας των φύλων. Το Σλοβενικό και Εστονικό Κοινοβούλιο το δοκιμάζουν, το ε, συζητούμε και με το ελληνικό, ώστε να καταγράφονται κάποια στοιχεία όπως η παρενόχληση σεξουαλική. Αλλά είναι στοιχεία στα οποία βασιζόμαστε για να καταγράψουμε αυτούς τους χάρτες ισορροπίας εξουσίας. Γιατί όπως λέτε και εσείς δεν μπορούμε απλά να παρατηρούμε αυτά τα φαινόμενα χωρίς να αναλαμβάνουμε καμία δράση. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Λάνμπεκ για την παρουσίαση, για τη συνεργασία. Θα τα ξαναπούμε 21 Νοεμβρίου όπου θα έχουμε τη συνάντηση της Επιτροπής μας με μέλη των Εθνικών Κοινοβουλίων και εσείς θα παρουσιάσετε τον δείκτη για την βία κατά των γυναικών. Σας ευχαριστώ.